Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω να καλωσορίσω τον κύριο Βίλαν επίσης ε, της Γενικής Διεύθυνσης Connect και τον κύριο Κάρτσο Μπλοκ ή κάπως έτσι τέλος πάντων Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση από πλευρά της Επιτροπής τη αξιολόγηση αντικτύπου του κανονισμού του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες. Θα γίνει μια εισαγωγή, το πολύ 15 λεπτών, από τον κύριο Βίλαμ. Θα ακούσουμε μια πολύ σύντομη ε, παρουσίαση από πλευράς της κυρίας, του, από πλευράς της Μπερέκ, συγγνώμη, έχουμε στη διάθεσή μας ε, μία ώρα. Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έρθουν αργότερα στις 10 η ώρα και οι συνάδελφοι για να ψηφίσουμε. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα, να σας πω ότι θα προσπαθήσω να περιορίσω τον περισσότερο την παρουσίασή μου για να αφήσω και χρόνο για, ε, για τη συζήτηση. Οι στόχοι της πρότασης είναι γνωστοί ε, ήδη σε αυτό το επίπεδο, αλλά καλό θα ήταν να τους επαναλάβουμε έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι πώς καταλήξαμε σε αυτούς τους στόχους. Ε, καταρχάς, ο βασικός στόχος είναι η συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς που θα στηρίζεται στην ελευθερία των παρόχων αλλά και των καταναλωτών. Ε, εδώ τονίζουμε τον σταδιακό χαρακτήρα της ε, ενοποίησης της αγοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την βιομηχανία των δικτύων. Εμείς στην Κομισιό έχουμε φροντίσει ιδιαίτερα να στηριχθούμε στις υπάρχουσες δομές, δηλαδή στο σύνολο, το σύνολο των οδηγιών από το 2009 και ε, η νομοθεσία Μπέρε και η νομοθεσία Roaming έχουν παραμείνει ανέπαφες, αλλά ε, εστιάσαμε στην ε, δημιουργία πάνω σε αυτά τα θεμέλια, αν θέλετε. Ε, οι αρχές ανταγωνισμού, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε όλες τις νομοθεσίες, παραμένουν ε, ανέπαφες και αυτές ακέρες όσον αφορά την, τον κανονισμό της αγοράς. Ε, βέβαια χρειαζόμαστε με, πια, με πιο ενισχυμένη αν θέλετε δράση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το ανοιχτό ίντερνετ. Βέβαια πρέπει να αφήσουμε και ε, χώρο για καινοτομίες. Αυτό το οποίο θέλουμε επίσης ε, και γίνεται και κάποια συζήτηση για την οικονομική ενοποίηση του τομέα. Λοιπόν, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, οικονομίες κλίμακας και αυτές οι, οικονομίες αν θέλετε να περάσουν στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού χωρίς όμως να θίξουμε την αποτελεσματικότητα των, ε, να θίξουμε μάλλον τους αποτελεσματικούς ε, εταιρείες, αποτελεσματικές εταιρείες ανεξάρτητα του μεγέθους τους δηλαδή ακόμα και μικρής κλίμακας εταιρείες ε, είναι ευπρόζεκτες επίσης στην e θεωρεί ότι προτείνουμε τις ελάχιστες κυβερνητικές αλλαγές και, και για όσον αφορά τον Μπάρεκ, αλλά και για το Σπέκτρουμ και, για τις... και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ε, ενιαία ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η Επιτροπή θα πρέπει να ξέρει ότι πρόκειται για μία πρόταση η οποία είχε μία πολύ σύντομη περίοδο κοίησης σε σχέση με τα συνήθη. Ε, ξεκίνησε με βάση τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο του Μαρτίου όμως κάναμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο για να υποφεληθούμε από τις ε, ήδη υπάρχουσες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει ας πούμε για το Open Internet ή ε, επίσης ε, να λάβουμε υπόψη μας τις δουλειά, τις, την εργασία που έχει κάνει η Μπέρεκ για τις εγκρίσεις παραδείγματος χάρη Εποφεληθήκαμε από μια ευρύτερη διαδικασία όπου συμμετείχαν ε, οι ενδιαφερόμενοι ε, και ε, πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, CEOs από, μεγάλη, από διάφορες εταιρείες. Υπάρχει ένας διάλογος, δηλαδή ο οποίος ακόμα βρίσκεται εν εξελίξη. Για το, επίσης στο Radio Spectrum στην ομάδα του Radio Spectrum ε, επίσης ε, Επομένως, πρόκειται για μία πρόταση η οποία έχει φτάσει στους νομοθέτες Ε, με κάποια επιταχυμένη διαδικασία αν θέλετε. Εμείς θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις ε, απόψεις όλων των ενδιαφορεμένων και ε, να τις ενσωματώσουμε στις προτάσεις που θα κάνουμε. Η κινητήρια δύναμη πίσω από τις προτάσεις μας είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον κατακαιρματισμό ο οποίος υπάρχει στις ε, ε, ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες παρά τους κύκλους αν θέλετε νομοθετικών πράξεων που προσπάθησαν να ρυθμίσουν τον τομέα αυτό. Καταρχάς έχουμε έναν κατακαιρματισμό όσον αφορά τις εγκρίσεις των εταιριών τηλεπικοινωνίας ε, εξαρτάται και από, τις, από τα κριτήρια και από τις προϋποθέσεις ε, που ε, διέπουν την ρυθμιστική προσέγγιση. Δεύτερον, βλέπουμε ότι υπάρχουν απτά δείγματα κατακαιρματισμού όσον αφορά τον, την κατανομή φάσματος για την ευρεία ζώνη. Υπάρχει και μία επιβράδυνση στις διαδικασίες, στο roll-out, ε, επίσης, ε, υπάρχει μία έλλειψη πανευρωπαϊκής πρόσβασης ε, σε ένα ιδεατό δίκτυο. Αυτό δυσκολεύει τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει και μια, ένας κατακαιρματισμός της αγοράς όσον αφορά την, ε, τα, τα συμφέροντα του τελικού καταναλωτή. Θα μπορούσα, αν θέλετε, να κάνω μία σύντομη επιλογή ε, αποδεικτικών στοιχείων και βλέπουμε ότι όσον αφορά τον, τις τιμές στον, στον τελικό χρήστη υπάρχουν ε, εμφανή δείγματα κατακαιρματισμού στα ανάμεσα στην χαμηλή, ε, στις χαμηλές τιμές, στο χαμηλό κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν θέλουμε ε, ε, μια ενισχυμένη ενιαία αγορά που θέλουμε να έχει μια σύγκληση των τιμών, δεν θέλουμε αυτή η σύγκληση των τιμών να είναι ο μέσος όρος των τιμών που παρουσιάζονται. Θέλουμε μια πιο, ε, μια πιο δυναμική αγορά όπου οι τιμές θα συγκλίνουν στις πιο ανταγωνιστικές, με τις τιμές των πιο ανταγωνιστικών χωρών, όπου το κόστος παροχής είναι χαμηλό, άρα η τιμή μονάδας είναι χαμηλή και για τον καταναλωτή, τελικό καταναλωτή. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση win-win. Επίσης, σε αυτή την επόμενη διαφάνεια, θα δείτε ότι υπάρχει μια διακύμανση και όσον αφορά ε, το, την κάλυψη 4G στην Ευρώπη και ποια είναι η σύγκριση με τις εταιρείες στην Αμερική. Κάποια εταιρεία καλύπτει το 90% εκεί το 90% του πληθυσμού, ενώ η, ο ευρωπαϊκός όρος χώρος δεν είναι ούτε καν 30%. Επίσης, και είναι μια φυσική συνέπεια αυτό ότι τα επίπεδα κεφαλουχικών δαπανών στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χαμηλότερα, αλλά υπάρχει και μια ε, τάση πιο ε, χαμηλή, αν θέλετε, στην Ευρώπη, λιγότερο έντονη στην Ευρώπη. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ε, έναν καλύτερο τρόπο πώς μετράμε την σχέση ανάμεσα στο ε, εγχώριο ΚΑΠ σε σχέση με τις πωλήσει. Εν κατακλείδη. Βλέπετε και μια γραφική παράσταση όπου αποδεικνύεται ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τα έσοδα όσον αφορά τη μεταφορά της φωνής, ε, ναι μεν είναι σημαντικά, αλλά μειώνονται σταδιακά. Βλέπετε τα τι κερδίζουμε από, την, από ένα τηλέφωνο, από μια κινητή, κινητή ε, επικοινωνία μέσω της φωνής και την κινητή επικοινωνία μέσω μετάδοσης δεδομένων. Τέλος πάντων, ε, Αυτά, αυτές είναι γνώσεις και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου όταν ε, μιλάμε για το roaming, για τις διεθνείς ε, επικοινωνίες. Ε, οι εταιρείε χρειάζονται επιχειρηματικά μοντέλα που να επιτρέψουν να πουλάνε δεδομένα και να μεταφέρουν δεδομένα και όχι φωνή που είναι κάτι το οποίο φθήνει. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε πρέπει να κάνουν αυτή την μετάβαση όλες οι εταιρείε, όχι μόνο αυτές που είναι στη δεξιά στην αριστερή πλευρά ε, της διαφάνειας, όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείε που βρίσκονται, που θέλουν να βρίσκονται σε αυτή την δυναμική αγορά και που αντιμετωπίζουν την πρόκληση από πλευράς μετάδοσης, από τη σκοπιά της μετάδοσης των δεδομένων, θα πρέπει να... Ε, επιμείνουν περισσότερο, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάποιο βάρος. Τώρα, ποιες είναι, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες στους οποίους πρέπει να εξετάσουμε. Ε, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα. Και οι δύο αυτές αρχές ε, είναι θεμελιώδους σημασία. Είναι αναπόφευκτο βέβαια σε μέτρα εσωτερικής αγοράς ε, ο περιορισμός του κατακαιρματισμού γίνεται με καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης υπογραμμίζουμε ότι δεν θέλουμε να εξαναγκάσουμε σε μια συγκέντρωση του ελέγχου κλάδο Απλώς θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε παρόχους ε, που θέλουν να αναπτυχθούν ε, να το κάνουν ε, χωρίς να προσκρούν σε περιτά εμπόδια. Το ίδιο ισχύει και για την επικουρικότητα. Φροντίσαμε να παρεμβαίνουμε μόνο που είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελεγμών και διακριτική ευχέρεια για τις ε, εθνικές αρχές, για τη διαχείριση του φάσματος και για τα έσοδα από αυτά. Οπότε γίνεται από τα κράτη-μέλη επιλογή των ε, προϊόντων, των εικονικών προϊόντων. Και με το καθεστώς αδειοδότης που προτείνουμε, έχουμε τον, ε, το, κοδεσπότη του κράτους ε, μέλους υποδοχής που είναι το αρμόδιο. Ε, ο ρυθμιστικός φορέας του κράτους μέλους υποδοχής είναι ο αρμόδιος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους, γενικούς και ειδικούς, ουσιαστικά εδώ σχηματοποιώ αυτά που είπα ήδη. Έχουμε κάποιες μορφές κατακαιρματισμού που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να διευκολύνουμε τους παρόχους των υπηρεσιών να λειτουργήσουν πιο απρόσκοπτα, διασυνοριακά και να υποφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε διάφορες επιλογές πολιτικής που διερευνούμε. Καταρχήν το βασικό σενάριο, το σενάριο αναφοράς, χωρίς καμία επιπλέον ε, επέμβαση. Μετά έχουμε την πρώτη επιλογή με συγκεκριμένες ε, μεμονωμένες παρεμβάσεις. Τη δεύτερη επιλογή συνδυασμένες κανονιστικέ προτάσεις με κάποια μέτρα και η τρίτη επιλογή είναι πιο φιλόδοξη και περιλαμβάνει και μια ενιαία ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή και για την ρύθμιση της αγοράς και για την διαχείριση του φάσματος. Καταλήξαμε τελικά στο συμπέρασμα ότι ναι μεν η τρίτη εναλλακτική είναι δελαστική, αλλά ω προ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογή της ε, δεν είναι τόσο εφικτή. Και ε, δεν είναι η συγκέντρωση αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά περισσότερο άμεσα αποτελέσματα. Γι' αυτό καταλήξαμε και διερευνώντας και εξετάζοντας εδελεχώς τις επιμέρους επιλογές, διαπιστώσαμε ότι μια δυναμική αγορά θα πρέπει να προσανατολίζεται και να αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές ε, των κρατών μελών. Έτσι έχουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε και 110 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το χρόνο, αλλά θα είχαμε και συνέπειες ε, σε άλλους τομείς που ε, επηρεάζονται από την ε, διασυνδεσιμότητα. Θέλουμε κυρίως καλύτερες επιλογές για τον καταναλωτή και αναβάθμιση ποιότητας. Φυσικά θα έχουμε και βραχυπρόθεσμο κόστος, γιατί σταδιακά θα εξαλειφθεί η περιαγωγή. Μέσω πρόθεσμα σε ό,τι αφορά τα, τις ε, υπεραστικές διεθνείς κλήσεις και έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα για το 2016 αλλά ακόμη και στην ε, χειρότερη περίπτωση <clears throat> της μη δράσης δηλαδή ε, το κόστος είναι ούτως ή άλλως χαμηλότερο από τα ωφέλη. Εδώ βλέπετε, δεν θα σας διαβάσω, την σύγκριση των διαφόρων ε, εναλλακτικών. Και εκεί προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στην έγκαιρη επέμβαση για βασικά σημεία. Γι' αυτό και ταχθήκαμε υπέρ της δεύτερης επιλογής και όχι υπέρ της τρίτης που ήταν πιο φιλόδοξη, αλλά χρονικά πιο χρονοβόρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίλαμ. Για τρία λεπτά θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρτσόπουλο από την Μπέρεκ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας εκφράσω τις απόψεις μου για την ε, πρόταση περί ενωμένης Υπήρου. Ε, έργο μας ε, είναι να προωθήσουμε τον συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντέρεκ λοιπόν είναι υπέρ μιας ισχυρής εναρμόνισης. Έχουμε στόχους στήριξης και ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς και δημιουργίας ε, βέλτιστων συνθήκων για καλύτερες επενδύσεις. Είμαστε ενήμεροι και έχουμε επίγνωση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και για τα αριθμιστικά κενά που υπάρχουν καθώς εξελίσσεται η αγορά. Όντως υπάρχουν πηγές ανάπτυξης που μπορούμε να διερευνήσουμε περαιτέρω και σίγουρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές της εποχής μας και της οικονομίας μας. Αυτό είναι κάτι που έχουμε επαναλάβει και στην ακρόαση για την έκθεση της κυρίας Τράουτμαν για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες. Δεν Συμμεριζόμαστε όμως αυτήν την ε, αρνητική εικόνα που υπάρχει για τις συνολικέ επιδόσεις των ε, τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Εμείς ε, στην ΕΝΤΕΡΕΚ ανησυχούμε ότι δεν διερευνώνται επαρκώς οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του κλάδου. Οι συνθήκες ε, και για τους επαρόχους και γενικότερα, το διοικητικό πλαίσιο, το φορολογικό καθεστώς, ε, η γραφειοκρατία, η ζήτηση της αγοράς κτλ. Ε, χάρη οικονομίας χρόνου δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις ε, τα επιμέρου στοιχεία τη πρόταση, Θα σα εκφράσω όμως ε, μόνο μερικέ ε, σκέψει σχετικά με την αξιολόγηση της ε, πρότασης αυτή. Όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, την τιμολόγηση και τι επιδόσει. Εδώ παρατηρούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΩΣΑ, οι Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα διείσδυση, όμω οι Ευρωπαίοι πολίτε απολαμβάνουν υψηλότερε ταχύτητε και χαμηλότερε τιμέ. Επίσης υπάρχουν ορισμένε ανησυχίε όσον αφορά τις διακυμάνσει των τιμών στην Ευρώπη. Έχω εδώ μια μελέτη από το Αμερικανικό Ερευνητικό ε, Ίδρυμα που συγκρίνει τις τιμές ε, στην Ευρώπη, στην ε, Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Και εκεί φαίνεται ότι για, τις, για την ευρυζωνικότητα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μόνο για την ευρυζωνικότητα και στα τριπλά πακέτα Παρατηρούνται διαφορές ως και τρεις φορές ε, παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη των δικτύων. Να σας πω ότι η ΠΕΡΕΚ στηρίζει απόλυτα τον ε, στόχο της ε, τόνωσης και της στήριξης των επενδύσεων μέσω ενός ε, ξεκάθαρου, σαφούς ε, και συντονισμένου πλαισίου σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν χρήσιμο εδώ να συζητήσουμε τις πιθανές εναλλακτικές ε, λύσεις για την καλύτερη ανάπτυξη των δικτύων. Όμως, να σας πω ότι οι επενδύσεις δεν έχουν παγώσει και δεν βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση στην Ευρώπη. Τα συστήματα και τα δίκτυα πρόσβασης αντίθετα αναπτύσσονται με ταχύτητα του ρυθμούς. Και αυτό θα οδηγήσει σε αποδοτικότερες επενδύσεις. Οι οπτικές ίνες αναπτύσσονται με εκπληκτική ταχύτητα στην Ευρώπη, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία για το FTTA και το FTTB σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, θα ολοκληρώσω την ε, παρέμβασή μου με ένα τελευταίο σχόλιο. Εμείς ε, θα θέλαμε και στην Ευρώπη να έχουμε παρόχους και υπηρεσίες όπως η Google και η Microsoft. Αυτό είναι το όνειρο των ε, καινοτόμων επιστημόνων μας και είναι κάτι που θα έπρεπε να σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει τώρα. Κύριε Τελκαστήγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, δεν εννοούσα εσάς, τον κύριο Τσίτσεστερ. Ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Είπατε στον εκπρόσωπο του Μπερέκο ότι είχε ένα πεντάλεπτο, εκτός κι αν δεν κατάλαβα καλά από τη διερμηνία. Αλλά τον κόψατε στα τέσσερα λεπτά. Υπάρχει λόγος, ενώ του δώσατε αρχικά πέντε. Ναι. Ναι, τον έκοψα γιατί του είχα, του είχα δώσει τρία λεπτά και όχι τέσσερα και όχι πέντε. Τρέ, τρία λεπτά έχει, τρία λεπτά έχει. Εγώ Λυπάμαι, αλλά εγώ άκουσα να λέτε πέντε. Μπορεί εγώ να παράκουσα. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να ήταν πρόβλημα να μην καταλάβατε καλά τη διερμηνία. Εν πάση περιπτώσει. Το αφήσαμε ούτω ή άλλω στον εκπρόσωπο του φορέα Μπερέ και να μιλήσει τέσσερα λεπτά. Η κυρία Πιλάρ, Δελκαστήγιο. Ε, δεν θυμάμαι τι άκουσα, δεν ξέρω τι άκουσα. Οπότε σας πιστεύω και εσάς κύριε Τσίτσετερ, αλλά πιστεύω και την πρόεδρό μας. Ο εκπρόσωπος ε, του Φορέα Μπερέκ είχε την ευκαιρία να μιλήσει, αλλά θα έχει και άλλες ευκαιρίες ο Φορέας αυτός να μας παρουσιάσει τις θέσεις του, γιατί έχει θεμελιώδη ρόλο και στις συζητήσεις μας καλό θα είναι να δίνουμε πάντα την ευκαιρία σε εκπρόσωπο του Μπέρεκ ε, να εκφέρει τη γνώμη του. Η μελέτη επιπτώσεων ε, έχει το ίδιο πρόβλημα με την ε, κανονιστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινοβουλευτική μας επιτροπή ήδη άσκησε κριτική στα θέματα αυτά με μεγαλύτερη ή ε, λιγότερη δρυμύτητα όταν ε, η αρμόδια επίτροπος μας παρουσίασε και μας ε, εξήγησε την πρόταση, είπαμε ότι όλα αυτά έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αναπόφευκτο, εξαιτία αυτής της πίεσης χρόνου, δημιουργήθηκαν διάφορες επιπλοκές που θα τις ε, ξεπερνούσαμε αν είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Το κείμενο είναι ογκώδες και περίπλοκο. Και από κανονιστική άποψη πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ πιο ευανάγνωστο, απλό, καθαρό κείμενο. Κάτι τέτοιο θα ελάφρυνε κάπως και το περιεχόμενο και θα έκανε το κείμενο πιο εύληπτο. Αλλά επαναλαμβάνω, το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ πιστικό. Και η μελέτη επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τις, δύο δυσκολ... από τις ίδιες δυσκολίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων, θα ήθελα να τονίσω τα εξή. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντώνιο Βίλαντ, μας είπε ότι αυτά τα θέματα συζητούνται εδώ και πολύ καιρό. Το θέμα του φάσματος, για παράδειγμα. Έχουμε ήδη κάνει εκτενείς συζητήσεις και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει πολλές μελέτες επιπτώσεων. Οπότε για το φάσμα και τον καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση του φάσματος και τον περιορισμό του κατακαιρματισμού είναι γνωστό θέμα εδώ και πολύ καιρό. Όταν όμως μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, αυτό είναι πραγματικά ένα νέο στοιχείο και γι' αυτό το στοιχείο χρειαζόμαστε μία πολύ πιο ε, διεξοδική μελέτη επιπτώσεων. Όπως μας είπε και εκπρόσωπος του Μπέρεκ, έχουμε διαφορετικά εθνικά αριθμιστικά πλαίσια και έχουμε και διαφορετικά φορολογικά πλαίσια στα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία που απαιτούν μια πραγματικά πολύ πιο ενδελεχή και ευρυθή μελέτη επιπτώσεων για να καταλήξουμε σε μια τέτοια πρωτοβουλία που είναι πραγματικά πρωτότυπη και καινοτόμα. Θα μπορούσα να επεκταθώ και σε άλλα σημεία, αλλά θα περιοριστώ σε αυτά προς το παρόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της αρμόδιας ε, καθήλη επιτροπής και το θέμα αυτό, ανέλαβε τη δέσμευση να προχωρήσει τη συζήτηση και να οριστικοποιήσει τη θέση του στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό το συμφώνησα εγώ ως εισηγήτρια με τους κοιόδης ηγητές της Επιτροπής, σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους ε, σκιώδης ηγητές ε, της Επιτροπής εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών, που είναι επίση συναρμόδια. Οπότε όλη αυτή η βιασύνη και το πιστικό χρονοδιάγραμμα μας προβλημάτισαν, αλλά πραγματικά επειδή υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην πρόταση, ε, θεωρήσαμε ότι αξίζει τον κόπο να τα προωθήσουμε και μάλιστα πριν την αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο που είναι και αναπόδραστη θα πρέπει να γίνει τέτοια αναθεώρηση και μάλιστα ρηξικέλευτη αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο, γιατί πολλές από τις διατάξεις της νέας ε, ρύθμισης ε, θα έχουν αντίκτυπο και θα απαιτήσουν την αναθεώρηση της οδηγίας. Οπότε το 2016 και μετά όταν θα γίνει αυτή η αναθεώρηση θα φτάσουμε άνετα στο 2018 μέχρι να έχουμε ε, και νέα μέτρα και να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και είπα και τις προάλλες, δεν θυμάμαι πού, ε, ο κόσμος του διαδικτύου δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε παρόν. Έχει μόνο μέλλον. Οπότε πολλές φορές το μέλλον, το αύριο δεν περιμένει. Θα πρέπει ήδη από τώρα να λάβουμε τις αποφάσεις και για το μέλλον. Και από αυτή την άποψη κάποιες προτάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσε και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τηρήσει την υπόσχεσή του, τη δέσμευση και την ευθύνη του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πιλάρ. Ο κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βίλαν που ήρθε σήμερα. Ωστόσο, Αναφέρατε τις απόψεις ε, των ε, ενδιαφερομένων. Και θα ήθελα να μου το αναπτύξετε αυτό το σημείο, διότι δεν ε, συμφωνεί με αυτά που έχω εγώ ακούσει από τους διαφορούς ενδιαφερομένους φορείς κατά τη διάρκεια μιας προφορικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφορούσε το γιατί δεν διεξήχθηκαν διαβουλεύσεις. Τώρα, μιλήσατε για ελάχιστες αλλαγές στη διακυβέρνηση και προτείνεται και αυτήν την μεταφορά αρμοδιοτήτων προς κεντρικές υπηρεσίες. Επίσης, αναφερθήκατε στην αξιολόγηση των ε, πλεονεκτημάτων των μέτρων αυτών. Αναφερθήκατε στο ποσό των 110 δισεκατομμύριων ευρώ και θα ήθελα πραγματικά να μάθω πώς ε, φτάσατε σε αυτό το νούμερο, ποια μέθοδο ακολουθήσατε για να το υπολογίσετε. Επίσης, ε, θα ήθελα να διαφωνήσω με τις απόψεις σας για τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Ε, υπάρχει μια διαφορετική άποψη, η οποία λέει ότι οι τέσσερις σε μεγαλύτεροι υπάροχοι κατέχουν το 60% της αγοράς. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό με αυτά που λέτε εσείς. Επίσης, Λυπούμε για το γεγονό ε, ότι εσεί πιστεύετε ότι η επιλογή 2 είναι καλύτερη από την επιλογή 1. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάντα καλύτερο να αναπτύσσουμε τα υφιστάμενα συστήματα και του υφιστάμενου ε, θεσμού και να του δώσουμε μια ευκαιρία να επιτύχουν παρά ε, να νομοθετούμε πρόημα. Επίσης, αναρωτιέμαι γιατί τόση βιασύνη για να δημοσιεύσετε αυτό το συνονθήλευμα προτάσεων διότι πιστεύω πως ε, δεν καθιστά αυτό μία ε, σωστή αναθεώρηση του κανονισμού. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει τόση βιασύνη για μια αναθεώρηση του κανονισμού και σε περίπτωση που υπάρχουν, γιατί να πρέπει να αναθεωρηθεί όλος ο κανονισμός. Επίσης, Λυπάμαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει στην προφορική μου ερώτηση πριν από δύο εβδομάδες και σημείωσα ότι απάντησαν πως θα στείλουν μια γραπτή απάντηση και πραγματικά περιμένω να τη δω. Σύντομα, να σας ε, προειδοποιήσω όμως ότι πρόκειται να σας στείλω και άλλες ερωτήσεις στο μέλλον, διότι αυτά που άκουσα μέχρι τώρα δεν με έχουν ικανοποιήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σομπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δεν μπορέσαμε να, συμπληρω... να ακούσουμε παραπάνω από τους δύο μιλητές μας, διότι από ό,τι φάνηκε ότι υπάρχουν και κάποιες μικρές διαφορές στις απόψεις τους και θα ήθελα ο εκπρόσωπος του Μπέρεκ να συνεχίσει την ε, παρουσίασή του. Μιλήσατε για τον κατακαιρματισμό. Ε, τι διαπιστώνουμε όμως ότι γίνεται. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της Υπέθρου, από το Massif Central. Εκεί εκλέγομαι, ε, στη χώρα μου, τη Γαλλία. Και τι διαπιστώνουμε, ότι αυτός ο ψηφιακός για τον ψηφιακό κατακαιρματισμό, ούτως ή άλλως ε, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλοι τα ίδια καθήκοντα, μένα, στον πόλεμο, στην ειρήνη κτλ, αλλά στην ειρήνη δεν έχει η χώρα, όταν η χώρα πάει καλά δεν έχουμε ίδια δικαιώματα και ε, όσον αφορά την άνεση ας και την ευζοία των πολιτών εμείς ε, έχουμε πάντοτε μια καθυστέρηση 5-10 χρόνια δεν ξέρω πόσα θα είναι αλλά πάντοτε ε, μας εξυπηρετούν ε, καθυστερημένα με το νερό, με, την υγειονομική περίθαλψη με, την, με τους αυτοκινητοδρόμους με τα τρένα κτλ. Και σήμερα τώρα είναι η ψηφιακή επικοινωνία Επομένως δεν θα πρέπει να το δείτε ε, για τον, τον, πρέπει να δείτε με διαφορετικό τρόπο τον ψηφιακό καταγερματισμό και διαρωτώ με ε, ποια είναι η λογική της αγοράς, η λογική των αγορών που είναι η λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η Ευρώπη και τώρα βλέπουμε ότι αυτή η λογική έχει κάποια όρια. Δεν θέλω να την αμφισβητήσω μένα αλλά θα πρέπει να μην κάνουμε ένα patchwork ανάμεσα στο ή θα πρέπει μάλλον να κάνουμε ένα patchwork ανάμεσα στους, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξυπηρετούνται. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και όταν απορρίπτεται την εναλλακτική λύση 3 κάνετε, διαπράτετε ένα σοβαρό σφάλμα. Ο κατακαιρματισμός από τι προέρχεται. Προέρχεται από το γεγονός ότι οι διάφορες εθνικές αρχές, ο Μπέρεκ που συντονίζει, τι συντονίζει τελικά, οι εταιρείε μας λένε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί στόχοι ενώ η τιμολόγηση γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ποιο κάνει τα δίκτυα, κανείς δεν κάνει τα δίκτυα πέραν της λογικής της αγοράς. Επομένως εγώ θέτω το ερώτημα, πώς μπορούμε να έχουμε μια κάλυψη και να καθησυχάσουμε τους πολίτες που να έχουν εμπιστοσύνη στην Ήπειρό τους, διότι όλοι ξέρουν ότι η πρόσβαση στην, ε, στην, ε, στην, ε, στην ψηφιακή αγορά, στην, στους αυτοκινητοδρόμους και στους τρένους είναι ένα θέμα αρμοδιότητας και επιτυχίας όλων μας. Ευχαριστώ κύριε Οντί. Προτείνω το εξής. Αφού δεν ακούστηκαν πολλές παρεμβάσεις και έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο πριν από, τις, από τα συμπεράσματα στον εκπρόσωπο του Μπέρεκ για να συμπληρώσει διότι, την παρέμβασή του, διότι άκουσα ότι κάποιοι συνάδελφοι είχαν και, κάποιοι, και κάποιες απορίες. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Μπέρεκ έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να επαναλάβω και να τονίσω προς όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής ΙΤΡΕ και, την και στην εισηγήτρια και τους και οδησηγητές ότι θα σας έχουμε στείλει ήδη... Ε, έχουμε στείλει ήδη απάντηση στη διαδικασία διαβούλευση που ξεκίνησε η κυρία Καστίγιο και μπορούμε να σας μοιράσουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτής. Εν συντομία τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατακαιρματισμό, η πάροχη κινητής ε, τηλεφωνίας ε, έχουν 221 ε, εκατομμύρια ουσιαστικά, οι δύο μεγαλύτεροι ε, πάροχοι έχουν συνδρομητές πολύ περισσότερους από ότι οι αντίστοιχοι μεγάλοι πάροχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχουν και ένα εθνικό αποτύπωμα, οπότε δεν ξέρουμε τι ε, ωφέλη θα έχουν ε, σε ό,τι φορά την οικονομία κλίμακος ε, και κατά πόσο μπορέσουν να μεγαλώσουν το αποτύπωμά τους, μια και το αποτύπωμα αυτό συνδέεται κυρίως με εθνικά δίκτυα. Ούτε γνωρίζουμε παραδείγματα υπηρεσιών που λείπουν αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν στο μέλλον οι πάροχοι να προσφέρουν στην αγορά. Ίσως θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και τους δυνητικούς κινδύνους μιας παγιωμένης ή συγκεντρωμένης διαδικασίας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη θέση των μεμονωμένων παρόχων. Επίσης, αναφέρθηκε η ενιαία ευρωπαϊκή άδεια, ο φορέας μας έχει υποβάλει προτάσεις για την ελάφρυση του διοικητικού άχθους των ε, παρόχων που δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι οι Ευρωπαίοι πάροχοι που ε, εισέρχονται σε μία μορφή αγορά θα πρέπει να έχουν επίγνωση των διαφορετικών νομικών συστημάτων, των φορολογικών συστημάτων και των διαδικασιών αδειοδότησης. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να έχουμε πιο απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης. γιατί μια υπερβολικά βαρημένη γραφειοκρατική διαδικασία θα επιτείνει την έλλειψη ασφάλειας δικαίου που υπάρχει μερικέ φορέ εξαιτία τη πολυμορφία των νομικών συστημάτων. Όπω είπα και στην αρχή, μπορούμε ε, να σα μοιράσουμε την ε, παρουσίαση που κάναμε, την ανάλυση που έχουμε κάνει στον Μπερέκ, σε όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ. Κύριος Μπίλαντ. Πρόεδρε, ας ξεκινήσω καταρχάς ευχαριστώντας τον εκπρόσωπο του Μπέρεκ, γιατί Ούτως ή άλλως και οι δύο πιστεύουμε ότι στον τομέα των εγκρίσεων υπάρχει χώρος βελτίωσης. Μεν, αλλά συμφωνούμε ε, σε κάποια πράγματα. Θα ήθελα να θίξω εν συντομία ε, σε, σε ένα θέμα που έθιξε ο ίδιος και ο κύριος Τσίσεστερ για το, το υπάρχοντο επίπεδο κατακαιρματισμού. Εάν δείτε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι γενικότερα στην Ευρώπη το, ο αριθμός δεν είναι τόσο ενσωματωμένος όσο στις Ηνωμένε Πολιτείες, ολοκληρωμένος στις Ηνωμένε Πολιτείες. Επομένως δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Αλλά δεν θα πρέπει να ε, μετρήσουμε απλώς τον αριθμό των ε, συνδρομητών. Έστω και αν έχετε πολλούς ε, περισσότερους συνδρομητές κάτω από την ίδια στέγη, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι, οι συνθήκες ανταγωνισμού από τις οποίες αποφελούνται. Και εδώ η κατάσταση δεν είναι ίδια. Όσον αφορά την εμπειρία των συνδρομητών υπάρχει μαζική, μαζικός κατακαιρματισμός και αυτό οφείλεται ίσως ε, και στις ε, κανονιστικές συνθήκες, ε, στην ποικιλία αν θέλετε, στα επίπεδα ανταγωνισμού, στις διάφορες, σε επίπεδα αρμοδιοτήτων συγγνώμη, σε διάφορες εθνικές αγορές, αλλά και συνθήκες στην αγορά ε, μέσω των ε, οποίων χορηγείται το φάσμα. Βέβαια, πρέπει να εξετάσουμε την καρδιά του προβλήματος. Πρόβλημα έτσι όπως ακριβώς το έχουμε εντοπίσει. Απ' την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να θεωρήσουμε σαν προϋπόθεση ότι αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα είναι αυτά, τα αυτό το οποίο θα πρέπει να ισχύσει δεν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εθνικών αγορών η ιδανική. Δεν ε, αν δούμε τι γίνεται στις, ε, στις άλλες, σε όλες τις χώρες, ε, τα εθνικά δίκτυα, Μάλτα, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία τέλος πάντων, σίγουρα αυτά τα εθνικά δίκτυα δεν είναι τα ιδανικά, δεν είναι τα βέλτιστα. Βέβαια, οι μεγάλες εταιρείες προφανώς εποφελούνται από καλύτερες συνθήκες το θέμα των ε, προνομίων, των κερδών, των, οφέ, ε, ε, του όφελου, του ωφέλους. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει και η έκθεση ΑΚΟΕΣ που είναι ένα κομμάτι των προτάσεών μας και εκεί γίνεται μια συντηρητική εκτίμηση του κέρδους που μπορούμε να έχουμε. Τι λέμε εκεί, ότι οι διάφορες ευρωπαϊκές αγορές θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες, βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικές. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι προς όφελος του ανταγωνισμού, διότι θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά έτσι ώστε η, ο τομέας να ε, προσανατολιστεί σε πιο βιώσιμα ε, μοντέλα που ε, θα στηρίζονται στα δεδομένα ενώ γιατί η δουλειά μας είναι να, πληρώσουμε, να πουλήσουμε συγγνώμη, σαν περισσότερα δεδομένα στον τελικό καταναλωτή. Εμείς ε, είδαμε τα θετικά, το θετικό αντίκτυπο σε κάποιες ε, εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Αγορά. Η ερώτηση του κυρίου Οντίο αναφορά το τιμολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι είναι, συγγνώμη, όχι, αφορά το κατακαιρματισμό. Ε, υπάρχουν, ε, ένα, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία βοηθούν. Στην ε, πρόταση αυτή εδώ είναι το ένα. Όσον αφορά το φάσμα, προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη να μπορούν να ορίσουν ε, προϋποθέσεις εθνικής κάλυψης έτσι ώστε το, η, η κατανομή του φάσματος να είναι ένας μηχανισμός για την ασύρματη κάλυψη και των πλέον απομακρυσμένων περιοχών και ξέρουμε ότι το ασύρματο για την οικονομία του δικτύου θα είναι η πιο αποτελεσματική τεχνολογία και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ε, και ένα άλλο στοιχείο είναι οι προτάσεις ε, της Κομισιόν για την μείωση ε, του κόστους ανάπτυξης ε, της ευρυζωνικής επικοινωνίας. Μιλάμε για περιοχές που η αγορά δεν θα προσπαθήσει να καλύψει σαν μια αντιμετώπιση του status quo. Τώρα, όσον αφορά την διαβούλευση που ανέφερε ο κύριος Τσίτσεσεν, Προφανώς δεν έγινε 12, ε, μια διαβούλευση 12 εβδομάδων, αλλά διαπιστώσαμε και από την δική μας γνώση του τομέα, αλλά και από τις συνεχείς επαφές που είχαμε, και με την επαφή που είχαμε και με, τον Μπέρεκα στέλος Ιουνίου και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όχι, και για να μην πω και την συζήτηση η οποία ξεκίνησε από, με βάση προηγούμενες εκδοχές που δημοσιεύθηκαν, ε, μπορέσαμε να κάνουμε σημαντικές προσαρμογές ε, όσον αφορά τις ε, θέσεις και τις απόψεις των ενδιαφερομένων. Δεν με εξέπληξαν πολλά από αυτά τα οποία άκουσα μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου από τους ενδιαφερομένους, διότι ούτως ή άλλως ε, τα είχαμε λάβει υπόψη μας. Βέβαια δεν ικανοποίησαμε τους πάντες, αλλά αν μη, τι άλλο τουλάχιστον ξέραμε τι θέλανε οι πάντες. Και μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες. Προφανώς η, η, η νομοθεσία από μόνη της δεν ε, βοηθάει την υγεία ή την ε, διατήρηση του τομέα ενός τομέα. Η πρότασή μας ε, προφανώς δεν επηρεάζει την δημοσιονομική θέση, όσον η πρόταση ε, για τις εγκρίσεις δεν ε, θίγει κάτι τέτοιο, διότι ούτως ή άλλως δεν θίγεται η δημοσιονομική πολιτική, η εφορολογία ούτως ή άλλως από μια τέτοια πρόταση. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα διακύμανσης, τα οποία δεν εξηγούνται απλά από εξωγενείς παράγοντες κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, ε, περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά το 2008 ή από το 2010 όταν ε, η κρίση για το εθνικό χρέος έγινε πολύ πιο έντονη και εμφανής. Πάντως τα, μέχρι πρόσφατα σε γενικές γραμμές η πολιτική μας δεν διέφερε πολύ από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα δεν θα δείτε, ε, δεν θα βρείτε δηλαδή αν θέλετε εκεί τους λόγους για την κατάσταση. Ωραία λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει η Πιλάρ. Σε αυτή τη φάση της συζήτησης ε, τι άλλο να πω. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Βίλαντ που μας κάνατε την παρουσίαση και ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο του Μπέρεκ μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία της ε, συζήτησης ε, στην Επιτροπή μας. Θα έχουμε και στο μέλλον πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πιλάρ. Ευχαριστώ τον κύριο Βουίλιαν και τον εκπρόσωπο του Μπέρεκ. Ε, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εργασίας μας για το, τους κανονισμούς για την τηλεπικοινωνία. Ευχαριστούμε τους φιλοξενούμενους μας, τους προσκαλεσμένους, τους προσκεκλημένους μας και προχωράμε στην ε, ψηφοφορία. Ωραία. Είμαστε παρόντες όλοι. Παρακαλώ καθίστε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα είναι η έκθεση Proust για το CARS 2020. Πριν όμως περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, για να ελέγξουμε το μηχάνημα. Άρχεται ψηφοφορία, παραλαμβάνω. Τέλος της ψηφοφορίας. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Ξεκινάμε τώρα. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία... Προφορική τροπολογία, συγγνώμη λέει Προφορική τροπολογία 21, ποιο είναι υπέρ. Ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 40 υπέρ 3 κατά. Τροπολογία 22 τώρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, τροπολογία 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, λέει πρόεδρο υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7, υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 39, πρώτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, 39, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 40, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 και 49 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 50 και 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 και 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 98, δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 102, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασ... Ε, τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 15 υπέρ κατά εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται, 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 126 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Στην βασική πρόταση 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 148 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία συμβασική πρόταση 19 εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150-151 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτονται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20, συμβασική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Απολογία 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 164 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 και 166 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187-188 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Θα περάσουμε πολλές τροπολογίες. Τροπολογία 22. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ιδεολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ανοιχτή ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. 37 υπέρ 4, 5 ε, κατά και 4 αποχές. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Σέντο ή Αλαμπάρ. Για τον Μπέρεκ. Λοιπόν, ε, τροπολογία 21, ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την τροπολογία 38 της κυρίας Τρότμαν ε, θα ήθελα να παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία. Είδα ότι στην, ε, στο κατάλογο των ψηφοφοριών υπάρχει αυτή η προφορική ε, τροπολογία με την σύμφωνη γνώμη της κυρίας Στικάου, η οποία δυστυχώς δεν είναι παρούσα. Ε, δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Ε, όλοι την έχετε μπροστά σας. Ε, καλό τους συναδέλφους να την ε, υποστηρίξουν. Συμφωνείτε, άρα την, ψηφίζουμε τροπολογία 38 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40, D, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44D και 45D υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 50D και 51D υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική πρόταση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 61D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, από κοινού οι τροπολογίε 1, 2, 3, 4 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 6 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογίες 14D και 15D υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 17D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, για, την, ε, για ε, ε, το budget 1 υπέρ κατά εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει, ε, ξεκινάμε. Πέρας ψηφοφορίας. 45 ψήφισαν, 44 υπέρ, 1 κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία της ε, Vicky Ford, την έκθεση Vicky Ford. για την έκθεση εφαρμογής του 2013 ανάπτυξη εφαρμογής τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε όμως, να ελέγξουμε λίγο την, ε, την, ε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το 25 ηλεκτρονικά. Πέρες ψηφοφορίας 35 υπέρ 7 από 7 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Όχι, συμβαστική πρόταση 2, υπέρ. Συμβαστική πρόταση 2. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, μάλλον συμβαστική πρόταση 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51. 51. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 και 57 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία της ημέρας, που είναι μία ενιαία ψηφοφορία, αλλά σε δύο προφορικές ερωτήσεις, μία απευθύνεται στο Συμβούλιο και η άλλη στην Κομισιόν, για το ΡΕΜΕΚ. Ψηφίζουμε. Για την έκθεση Ρέμεκ φαντάζομαι. Ναι. Πέρα τη φιβορίας. 44 υπέρ, μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους. Ολοκληρώσαμε την, τις ψηφοφορίες πολύ συγκροτημένα και γρήγορα. Grazie a tutti. Allora chi deve Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, όσοι θέλετε να ε, φύγετε από την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνετε χωρίς ε, φασαρία. Έχετε τρία λεπτά για να καταλήψετε την αίθουσα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να καθίσουν. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους, μια και η κυρία Άντερσον ε, έρχεται, μήπως θα μπορούσαμε, για να μην χάνουμε ε, και το χρόνο μας, να ασχοληθούμε τα δύο τελευταία σημεία της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο κύριος Τοντενόφσκι, το Σενόφσκι είναι έτοιμος, θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση για, τις, ε, για, τον, ε, για τον τριμερή διάλογο που τον αφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τριμερής διάλογος για το ευρυζωνικό ίντερνετ στο πρόγραμμα CIF θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα. Θα είναι η δεύτερη συνεδρίασή μας. Ε, έχει πολλά τεχνικά σημεία, πολλές τεχνικές πτυχές και δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τρεις ακόμη εκκρεμότητε και είμαι αισιόδοξο. Ευελπιστώ ότι θα τις διεκπαιρώσουμε στην απογευματινή μας συνάντηση. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συγκλίνουμε τις απόψεις μας και να φτάσουμε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Γιατί ήταν μήνες οι συζητήσεις για το θέμα αυτό Εξαιτία ε, της αλλαγής και του προϋπολογισμού, κάτι που επηρέασε τις συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά το ευρυζωνικό διαδίκτυο, μειώθηκε το κονδύλιο από τα 10 δις στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ Μεγάλη περικοπή, δρακόντια. Πάντως ελπίζω ότι σήμερα το βράδυ με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε τον τριμερή διάλογο. Βέβαια δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα, αλλά όπως σας είπα είμαι αισιόδοξο γιατί όλοι δείξαμε διαλλακτικότητα και πνεύμα συνεργασίας και αναζήτηση κοινών σημείων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στη νομική μας υπηρεσία και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Βιομηχανίας και Έρευνας. Επαναλαμβάνω, είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας θα στεφθούν με επιτυχία. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας έγινε πριν από πολύ καιρό, μήνες ολόκληρους. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μετά και τη σημερινή βραδινή συνάντηση να καταφέρουμε να διαβάσουμε το ζήτημα στην Ολομέλεια. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο. Ε, θα ήθελα να σας δώσω και μια πληροφορία προς όλους τους συναδέλφους ε, και προς την Κομισιό για τις αποφάσεις των συντονιστών που συνεδρίασαν χθες το απόγευμα. Καταρχάς, όσον αφορά την ε, ομάδα επαφής ΑΣΕΡ ε, αποφασίστηκε να ζητήσουμε και από άλλους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να κάνουν μια ετήσια συνεδρίαση με την ομάδα επαφής και για την ε, Επιτροπή Ήτρε να υπάρχει μια ετήσια επίσκεψη για την παρουσίαση της έκθεσης ΑΣΕΡ. Αυτά για το θέμα Άσερ. Επίσης, αποφασίστηκε να υπάρξει μία δημόσια ακρόαση για το πρόγραμμα το οποίο για τον ΕΡ 300 ε, η πρόταση που έγινε 9 Οκτωβρίου έγινε δεκτή επίσης ε, στο 1D για το σύστημα κατανομής ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έκθεση ε, δόθη στο ΕΛΚ. Επίσης, μία πληροφορία για το ταξίδι. μιας αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ήτρε από τις 26 έως 30 Αυγούστου. Στο ταξίδι αυτό, εκτός από μένα, πήραν μέρος η κυρία Ντεκαστίγιο, κύριος Λάγκε από το ΕΛΚΑ, Χέρτζογκ, Ρέσμαν και Ματίας, όπως επίσης και από πλευράς γραμματείας, Μπάγερ και Λέσνιακ. Η αντιπροσωπεία που προεδρεύω, που, της οποίας ε, προείδρευα εγώ έμεινε 1,5 μέρα στην Κορέα και την ημέρα αυτή είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε την εταιρεία Samsung και να κατανοήσουμε την ε, ε, σημασία, την μεγάλη σημασία που έχει αυτή η εταιρεία και για την Κορία, Κορέα καταρχάς, αλλά και για τον δυτικό κόσμο εν γέννη. Μετά συναντήσαμε και την ε, ε, τον, ε, την Επιτροπή της, την, ε, της Περιφερειακής Κυβέρνησης που ασχολείται με το εμπόριο. Εκπροσ, συναντήσαμε και προσώπους του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου και ε, είδαμε ακριβώς ποια είναι, ποιες είναι οι συνέπειες της νέας πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μετά συναντήσαμε και τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Εμπορίου της Κορέας για να δούμε ε, πώς εξελίσσεται το διεθνές, πώς επηρεάζεται το διεθνές εμπόριο από την, ε, από την συμφωνία ε, που υπογράφει πρόσφατα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κορέα. Μετά πήγαμε στην Ιαπωνία, όπου είχαμε πάρα πολλές επαφές αυτές τις δύο μέρες που μείναμε στη χώρα αυτή. Συναντήσαμε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, ε, της ε, ομάδας ε, έρευνας μιας επιτροπής ανεξάρτητης που εξέτασε το ατύχημα της Φουκουσίμα να δουν, δηλαδή εξετάζουν ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα. Ο κύριος Τανάκα που ήδη έχει πάρει τον λόγο στην Επιτροπή μας για να μας μιλήσει για την ε, ενεργειακή ε, ασφάλεια, αν θέλετε, της Ιαπωνίας. Επίσης, ήταν εκεί. Επίσης, συναντήσαμε και, τον, ε, και τους εκπροσώπους από, το, από την Φουκουσίμα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ακριβώς. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπάρχουν ε, κοινά σημεία ανάμεσα ε, στο πρόγραμμα της Ιαπωνίας και τον ορίζοντα 2020 το δικό μας. Οι επαφές αυτές μας επέτρεψαν να δούμε ότι υπάρχουν πολλές συνεργασίες, δυνατότητες συνεργασίες ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, όχι μόνο όσον αφορά την έρευνα, αλλά και σε άλλους τομείς. Όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, ε, συναντήσαμε εκπροσώπους της νέας υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας που είναι σήμερα ανεξάρτητη. Συναντήσαμε και επισκεφτήκαμε το κέντρο ελέγχου το οποίο ασχολείται με τα επεισόδια αυτά, με τα ατυχήματα. Ε, είδαμε την, είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με τον πρώην Πρωθυπουργό Ναότο Καν, ο οποίος μας εξήγησε ε, ποια είναι η δική του άποψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τομέα αυτό. Δείξαμε μεγάλο ενδιαφέρον ε, για τα όσα συμβαίνουν και σαν ε, συμπέρασμα αυτού του ταξιδιού η αντιπροσωπεία της στην Κορέα και στην Ιαπωνία να σας πω ότι το ταξίδι αυτό θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλη την αντιπροσωπεία, διότι το πρόγραμμά μας ήταν γεμάτο συναντήσεις και ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο. Όσον αφορά τώρα ε, τη, ε, τους συναδέλφους που θέλουν να ενημερωθούν ε, περαιτέρω για την, την επίσκεψή μας, έχουμε φέρει και διάφορα έγγραφα μαζί μας τα οποία είναι στην διάθεσή σας, τα έχει η γραμματεία και εάν το θεωρείτε χρήσιμο μπορούμε να σας τα διαβιβάσουμε έτσι ώστε να διαμορφώσετε μια συγκεκριμένη ε, άποψη για, το όσα, για τα όσα κάναμε. Τώρα, εάν κάποιος συνάδελφος που συμμετείχε στο ταξίδι θέλει να πάρει το λόγο, αλλιώς μπορούμε να περάσουμε μάλλον να μπορούμε να επιστρέψουμε στην ημερήσια διάταξη. Α, επίσης να συμπληρώσω ότι υπάρχει και το σημείο της α, κυρίας Βαλεάν, εδώ μίλησε ε, ο κύριο, μια και μίλησε ο κύριος Σασονόφσκι, λοιπόν, ε, να μας μιλήσει η κυρία Βαλεάν για τον ε, τριμερή διάλογο που, μας, που, που παρακολουθεί. Και μετά θα επιστρέψουμε στην ημερησία διάταξη. Κυρία Βαλεάν. Ε, με συγχωρείτε, ρωτήστε για τον τριμερή διάλογο. Δεν κατάλαβα ακριβώ. Ή για το εικόλ. Κοιτάξτε, μια και είπαμε ότι θα συζητήσουμε πρώτα τα τελευταία δύο σημεία της ημερησίας διάταξης, ε, καλό θα είναι να μιλήσετε για τον τρίλογο. Για τον τρίλογο σας μίλησα εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον τριμερή διάλογο για την έκθεση για τα επενδυτικά έργα στι υποδομέ τη ενέργεια. Τον δεύτερο, γιατί είχαμε ήδη έναν πρώτο τριμερή διάλογο. Ο κανονισμός αυτός για την τροποποίηση των επενδυτικών έργων στις ενεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπευλήθη στο Κοινοβούλιο, όπως είπα, δεύτερη φορά, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακύρωσε τον ε, κανονισμό του 2009 ε, όταν το Κοινοβούλιο με επιτυχία αμφισβήτησε την νομική βάση. Το πεδίο εφαρμογή είναι παρόμοιο με τον ε, παλαιότερο κανονισμό. Πολλές όμως τροπολογίες που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2010 συμπεριλήφθηκαν στο νέο κανονισμό. Μπορώ να σας αναφέρω ότι τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που δημοσιεύτηκαν πριν από δύο εβδομάδες είναι πολύ θετικά. Όσον αφορά ε, τώρα ε, τι ζητούμε. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αποφύγει τον επιπλέον φόρτο για, ε, για τα νέα έργα. Ζητούμε νέα, νέους κανόνες εμπιστευτικότητας, Ευκρινίστηκε το πεδίο εφαρμογή για τα έργα ενεργειακών υποδομών στον τομέα του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, λιγνίτη και την εμόλυνση καθώς και έργα που σχετίζονται με παραγωγή βιοκαυσίμων και δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας επίσης συμπεριλήφθηκε. Επίσης, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στην αναθεώρηση του 2016 μία πιθανότητα να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε την εξόριξη φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα, πεπιεσμένου φυσικού αερίου και να συμπεριληφθούν όρια για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση των ορίων αυτών. Αυτό το τελευταίο πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρεται στην ε, τοπική παραγωγή από μικρότερες μονάδες, κάτι το οποίο ε, αποκτά λιώνα και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μέλλον πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα των δεδομένων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Επίσης, καθορίσαμε σαφέστερα την ε, χρήση των δεδομένων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέσο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με αποτελεσματικότητα και όχι μόνο χάρη συλλογή δεδομένων. Στόχος είναι να εντοπίσουμε κενά στον ενεργειακό εφοδιασμό και εμπόδια που αφορούν τις επενδύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αναγκαίες και κατάλληλες πολιτικές στην ενεργειακή αγορά. Συνδυασμένο τώρα το, πρόγραμμα, το κανονισμός αυτός με την ε, διευκολύνση συνδέοντας Ευρώ, την Ευρώπη, σκοπός είναι να συνδέσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το υφιστάμενο δίκτυο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βαλεάν για την ενημέρωση αυτή όσον αφορά την εξέλιξη των τριμερών διαλόγων επί του θέματος της και περνάμε τώρα στην δική σας έκθεση βέβαια για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος e σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόφαση για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού πανευρωπαϊκού συστήματος e-call, όπως γνωρίζετε, συνοδεύεται με έναν κανονισμό για την ανάπτυξη του e-call στα οχήματα. Είμαι επίσης συγγήτρια για, για την έκθεση αυτή, αλλά με αυτή θα ασχοληθούμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Τώρα, η πρώτη πρόταση που εξετάσουμε σήμερα είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση για όλα τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν το, την, ε, τις αναγκαίες υποδομές για το σύστημα e-call, δηλαδή κέντρα λήψη κλήσεων έκτακτη ανάγκη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, η συνέχεια και ίσω καλή λειτουργία του ε, διαλειτουργικού πανευρωπαϊκού συστήματος ε, e-call. Καλωσορίζω την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι το σύστημα αυτό e-call στα οχήματα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των ε, θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και των ε, σοβαρών τραυματισμών. Συνειδητοποιούμε κοιτάζοντας τα στατιστικά στοιχεία ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. το 2012 είχαμε περίπου 20.000 ε, θύματα τροχαίων και πάνω από 2,5 εκατομμύρια τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα. Επίσης αυτό επιφέρει και οικονομικό φόρτο ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο το σύστημα e-call μπορεί να μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης των υπηρεσιών ε, εκτάκτης ανάγκης κατά 10 περίπου λεπτά, ειδοποιώντας τις ε, υπηρεσίες εκτάκτης ανάγκης άμεσα, ακόμα και αν ο οδηγός ή οι επιβάτες ε, δεν είναι σε θέση να καλέσουν. Οι συσκευές αυτές επιταχύνουν την άφηξη των υπηρεσιών εκτακτής ανάγκης κατά 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στην Ήπεθρο ως εισηγήτρια στηρίζω απόλυτα την πρόταση και υπέβαλα ελάχιστες τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία που υπέβαλα αφορά τα ε, δεδομένα ανάπτυξης για την 1η Οκτωβρίου 2015. Τα δεδομένα αυτά μου φαίνονται αρκετά φιλόδοξα από μεριά ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όντω οι τεχνικέ ε, προδιαγραφές, τα τεχνικά πρότυπα και η προσαρμογή χρειάζεται να ε, οριστούν μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση και πιστεύω ότι το 2015 είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πω τα κράτη-μέλη δεν θα προλάβουν να δημιουργήσουν τι αναγκαίε υποδομέ και να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μία αναβολή 9 μηνών που θα φτάσει το 2016 δηλαδή. Δεύτερον, θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη που ε, υπάρχει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι ε, διαθέσιμες σε όλους και όχι μόνο στους ε, οδηγούς οχημάτων. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζήτησε μία αξιόπιστη μέθοδο εντοπισμού μέσω κλήσεων υποβάλαμε μια γραπτή δήλωση ε, σε ψήφισμα το 2011, σύμφωνα με και με μια κοινοβουλευτική ερώτηση τον Μάιο του 2013. δυστυχώ και παρά την ε, διαθέσιμη τεχνολογία δεν έχει γίνει καμία πρόταση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάπτυξη του συστήματος e-call επιβεβαιώνει ότι ο εντοπισμό ε, και τα δεδομένα GNSS μπορούν να ανακτηθούν αποτελεσματικά μέσω των δικτύων κινητή τηλεφωνία και από άλλου ε, παρόχου. Δεν αμφισβητούμε την σημασία που έχει το e-call, όμως μέχρι τώρα ανέρχεται στο 1,7% των αιτήσεων κλήσεων ε, σε υπηρεσίε έκτακτη ανάγκη. και πιστεύουμε πως αυτό είναι ε, μια πολύ άσχημη συγκυρία ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τοχαίου τριχήματος. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας εντοπισμού, γεωγραφικού εντοπισμού μέσω των ε, δικτύων κινητής ε, τηλεφωνίας. Αυτό το σύστημα θα διασφαλίσει την εμεχιστοποίηση των ε, κοινωνικών ωφελών που θα έχει η χρήση γεωγραφικού εντοπισμού. Υπολογίζεται ότι πάνω από 5 δισεκατομμύρια κλήσεις e-call θα γίνονται κάθε χρόνο σε σύνολο 320 εκατομμύριων κλήσεων e-call. Στόχο είναι να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι οδηγοί που διαθέτουν το σύστημα αυτό στα οχήματά τους από το e-call και από τον γεωγραφικό εντοπισμό. Και χαίρομαι σε αυτό το σημείο πάρα πολύ που υπευλήθη μία παρόμοια τροπολογία στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή ΙΝΚΟ πιστεύω πως πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω επίσης ειλικρινά ότι ε, το Κοινοβούλιο θα καταφέρει να υψώσει το ανάστημά του στο ε, ζήτημα αυτό όπως και στο παρελθόν και θα στηρίξει την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο συνάδελφος Μπέλεκ. Σας ευχαριστώ. Όντως, θα συζητήσουμε τον κανονισμό σε ό,τι αφορά το, την πιστοποίηση και των οχημάτων με τη συμπερίληψη του, της συσκευής για το e-call. Είναι από τα πιο ευαίσθητα σημεία και, και πιο, το πιο χρονοβόρο. Η κυρία Βαλεάν ασχολείται με το PSAP, δηλαδή το Κέντρο Λήψης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης. Θα ήθελα απλώ να πω συντομία πως συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια της ηγήτριας. Ήδη μας υπενθύμησε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το περσινό του Ιουλίου και τη γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα περισσότερα στοιχεία ε, έχουν συμπεριληφθεί ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυστυχώς όχι όλα. Γι' αυτό και με τις ε, τροπολογίες που προτείνει η Συγήτρια ελπίζω να γίνουν και αυτές οι διορθώσεις. Οι τροπολογίες της είναι Σωστέ οδεύουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά είναι σημαντικό τα κράτη-μέρη να λάβουν μέτρα ήδη από τώρα, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ε, αναπτύξουν τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές και να συμπεριλάβουν ε, τα e-call προκειμένου τα κέντρα λήψη κλήσεων να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες κλήσεις. Μας ανέφερα τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία η κυρία Βαλεάνα, μην τα επαναλάβω. Είναι τεράστιο το πλεονέκτημα της εγκατάστασης ε, ε, του συστήματος e-call στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Επιτροπή Μεταφορών πρότεινε να εμείνουμε στην 1η Οκτωβρίου του 2015 την αρχική ημερομηνία για τα εγγένεια αυτού του συστήματος. Μακάρι να ήταν εφικτό αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι πολύ σύντομα, ούτε δύο χρόνια. Διαρωτόμαστε λοιπόν αν είναι εφικτό για όλα τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν αυτό το σύστημα e-call στα οχήματά τους ε, σε λιγότερο από δύο χρόνια, όπως σας είπα. Μακάρι να ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά συμφωνώ και με την πρώτη κυρία Βαλεά να δώσουμε στο Εναυτοκινητοβιομηχανία, στα κράτη-μέλη, στα κέντρα λήψης κλήσεων εκτάκτου ανάγκης, ένα επιπλέον οκτάμινο εννιάμινο και να παρατείνουμε την προθεσμία. Πολλά πιλωτικά προγράμματα και εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται τα προγράμματα χείρο 1 και 2 για παράδειγμα. Ε, ελπίζω να είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μας ενημερώσει για την διάμεση κατάσταση και την έκθεση πρόοδου για τα προγράμματα αυτά, για να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε πιο εμπεριστατωμένα μια απόφαση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση της για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος ε, γεωγραφικής τοποθέτησης. Ε, δηλαδή, να μην έχουμε μόνο εντοπισμό των ε, συστήματος e-call, αλλά να γίνεται εντοπισμό γεωγραφική θέση για οποιαδήποτε κλίση που αποστέλλεται στη γραμμή εκτάκτου ανάγκη 112. Γιατί οποιαδήποτε κλίση μπορεί να εντοπιστεί γεωγραφικά χάρη στο GNSS. Αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, φυσικά κανένα δεν θα ήταν κατά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Όπω είπε η κυρία Βαλεάν, τα e-call από αυτοκίνητα σε τροχέα είναι λιγότερο από 2% του συνόλου των κλήσεων εκτάκτου ανάγκης, ε, ιδιαίτερα από τις υπηρεσίες του 112. Οπότε θα ήταν ε, ε, ευάρεστο να διευρύνουμε την τεχνολογία εντοπισμού σε όλες τις κλήσεις ε, και ε, τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης μέτρου του 112 χάρη στη χρήση του GNSS και όχι μόνο του e-call. Ευχαριστώ κύριο Στοσενόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το σύστημα είναι πολύ χρήσιμο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το σύστημα GNSS ε, και τον εντοπισμό της θέσης. Είναι μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτενώς. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε μια σωστή διαδικασία και για τα θύματα αυτών των τροχιών ατυχημάτων, γιατί είναι πολύ εύθραυστη ε, και βάλω τη ψυχολογική τους κατάσταση και να μην δίνουμε την αίσθηση ότι κάποιος άλλος θα λαμβάνει αποφάσεις ερήμην τους. Είναι πολύ περίπλοκη αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την θέση των θυμάτων των τροχαίων. Όπως είπε η συγγετρία και ο προλαλής ε, το 2015 που είναι η προτινόμενη η ημερομηνία στόχος ε, είναι, παρά είναι νωρίς κατά τη γνώμη μας. Και επειδή είναι διαφορετικά τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της πρότασης για την ενσωμάτωση του σήματος e-call θα είναι πιο χρονοβόρα. Γιατί τα συστήματα κλήσεων εκτάκτου ανάγκη δεν είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιε υπηρεσίε επίση ε, είναι διαφορετικέ. Οι αρμόδιε υπηρεσίε που απαντούν σε τέτοιε κλήσει εκτάκτου ανάγκη. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ζωή και θανάτου η παράταση κατά ε, έστω και ένα χρόνο ή, λιγότερο που προτείνει η συγγήτρια. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να γενικευτεί η χρήση του συστήματος και φαντάζομαι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο η πλήρης εφαρμογή του εξαιτίας της πολυμορφίας ε, των εθνικών συστημάτων. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη και στον κλάδο για να εφαρμόσουν το σύστημα απρόσκοπτα. Επίσης, ό,τι αφορά την διαδικασία εντοπισμού, τη δυνατότητα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, θα ήθελα να πω, όλα τα αυτοπαντοποιημένα συστήματα διάσωσης ε, είναι πολύ ευαίσθητα. Γι' αυτό και τα κέντρα ε, λήψη των κλήσεων θα έχουν και κάποιε νομικές ευθύνε για την ε, κινητοποίηση των διαδικασιών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τις νομικές πτυχές. Θα πρέπει το σύστημα να είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Συμφωνώ με την ε, γνωμοδότηση γιατί πραγματικά είναι πολύ μεστή, αγγίζει όλα τα ευαίσθητα θέματα και τα τεχνικά είναι πολύ καλή έκθεση, αλλά θα πρέπει να είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο συνάδελφος κ. Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και κυρίως ε, σχετικά με τους ε, αυτοματισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, για τα ατυχήματα ε, τα δικά ατυχήματα μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε άμεσες πληροφορίες ε, όσον αφορά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, όσον αφορά την ε, τοποθεσία. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε βέβαια κάποιες ε, διαθέσιμες τεχνολογίες. Υπάρχουν όμως και άλλα ατυχήματα τα οποία δεν μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας αυτές τις βασικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Και πρόκειται για πληροφορίες που θα μπορούσαν να ε, διατίθενται από παρατηρητές, από παρόντες παρατηρητές, από αυτόπτες μάρτυρες στην, ε, στο ατύχημα. Και θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα, παραδείγματο χάρη, να υπάρξει μία πληροφορία και όσον αφορά την τοποθεσία και όσον αφορά τη σοβαρότητα μέσω ας πούμε της κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ε, βάσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες και όσον αφορά τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης αλλά και για τον τύπο του ατυχήματος και να έχουμε και μία πληροφόρηση ε, και για τη σοβαρότητα εκτός από τον γεωγραφικό εντοπισμό μάρτυρες ε, των ατυχημάτων θα μπορούσαν να έχουν την δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες σε έναν πραγματικό χρόνο όσον αφορά το ατύχημα. Διαφορετικό, διαφορετικές πληροφορίες από αυτές που δίνει η τροχέα παραδείγματος χάρη. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Θα είναι μια ε, μια application, ας πούμε, ένα application και στα smartphones. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Πρόντι. Δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Κομισιόν. Α, εδώ είναι, εδώ είναι. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έπρεπε να μιλήσω στην Επιτροπή Μεταφορών ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ε, γι' αυτό και δεν θα καταφέρω ενδεχομένω να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει που μου υποβλήθηκαν σήμερα. Προτείνω λοιπόν να σα απαντήσω γραπτό, σε όσε δεν θα μπορέσω να απαντήσω προφορικά. Τώρα, όσον αφορά τι ε, τροπολογίε τη πρόταση. Πιστεύω πως τουλάχιστον μία τροπολογία έχει σχέση με τα όσα άκουσα για το 112 και τα κινητά τηλέφωνα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Καταλαβαίνουμε τον στόχο των τροπολογιών αυτών, ότι δηλαδή θέλουν να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο υπηρεσιών είναι ακριβώς το ίδιο και για τους χρήστες του 112, ανεξάρτητα αν εκείνοι χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή το e-call στο αυτοκίνητό τους. Ωστόσο όμως θα είναι πολύ δύσκολο να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, διότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι διαφορετική. Άλλη τεχνολογία υπάρχει παράδειγμα στα κινητά τηλέφωνα με δυνατότητες ε, ε, δορυφορικής πλοήγησης όταν η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη. Άλλη δυνατότητα έχουν οι χρήστες όταν ε, καλούν το 112 σε εσωτερικούς χώρους όπου το σήμα δεν είναι καλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον στόχο των τροπολογιών αυτών. Πιστεύουμε ωστόσο ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισότητα στις, ε, στην παροχή υπηρεσιών. Επίσης να πω ότι ο αριθμός 112 είναι ένας παγκόσμιος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης και πιστεύω πως θα ε, πρέπει και τα κινητά τηλέφωνα να ακολουθήσουν το ίδιο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ, λέει η όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν την έκθεση και εμένα. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα σταθεί ενωμένο στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και εκτιμώ την στήριξή σας. Ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι δεν με εκπλήσει το επιχείρημά σα. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται εξάλλου εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζουμε όμως να υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί έτσι θα βρεθεί λύση. Αρκεί η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να συμφωνήσουν, γιατί οι εφαρμογές ε, και οι δυνατότητες υπάρχουν για να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. και σε αυτό το στάδιο μένει να το αποδεχτεί η Επιτροπή. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ελπίζω να καταλήξουμε σε θετικά συμπεράσματα για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βαλεάνα. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 5η 7 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησία διάταξης που αφορά το πρόγραμμα υποστήριξη για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος και γενικότερα για την παρακολούθηση των αντικειμένων στο διάστημα. Η κυρία Άντερς Ντότερ είναι άρρωστη, η συνάδελφός μας, ε, της ευχόμεθα περαστικά και ζήτησε ο συνάδελφος κύριος Τζόνσον να παρουσιάσει την έκθεσή της. Έχει το λόγο συνάδελφε. Ε, yes, ε, thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, απλώς θα διαβάσω τη δήλωση της Αμέλειας Ανταστότερ και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί Πρώτη φορά τη διαβάζω, πρίμα βίστα. Θα σας την παρουσιάσω όμως για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψε. Λέει λοιπόν η Αμέλεια, αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης για την ε, σύσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Επιτήρησης και Παρακολούθησης του Διαστήματος. Το σύστημα αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ικανότητας παρακολούθησης ε, του διαστήματος ε, και παρακολούθησης των ε, διαφόρων αντικειμένων ώστε να απεφευθεί ο κίνδυνος συγκρούσεων μεταξύ τεχνητών αντικειμένων, δορυφόρων ή θραυσμάτων από εκρήξεις στο διάστημα. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις παγκόσμιες προδιαγραφές και ο κλάδος και οι δημόσιες αρχές, γιατί όλοι εξαρτώμαστε από τις υποδομές στο διάστημα. Η πρόταση είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσουμε και μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των ε, δορυφόρων του γαλλία και του Κοπέρνικου. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να έχουμε μια τέτοια πρόταση που είναι άνευ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τις δεξιότητες των κρατών μελών προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στους χρήστες. Λέει λοιπόν η Αμέλη Αντερστότερ ότι προτείνω για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ε, μία συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και καταθέτω την τροπολογία 28 στο άρθρο 10 γιατί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι ο μόνος εγκεκριμένος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το SST και το SSA. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δεν μπορεί να ελέγξει το πρόγραμμα, θα πρέπει τουλάχιστον να συμβάλλει με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τους αισθητήρε 3α, 3.1α και εκεί θέλουμε ε, να διαγράψουμε την μνήμα υπαρχών των αισθητήρων, ώστε να αποφευθεί σύγχυση, ε, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στο σύστημα τους μελλοντικού αισθητήρε και αυτούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Ό,τι αφορά τη λειτουργία τώρα των υπηρεσιών, άρθρο 4, είναι πολύ καλή κατάταξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω να προσθέσουμε οποιασδήποτε συναφείς υπηρεσίες που κρίνει σκόπιμες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η ΕΣΑ και να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα για τις μελλοντικέ βελτιώσεις που θα προκύψουν από τις παρατηρήσεις των χρηστών ή των διαφόρων φορέων. Το πεδίο των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει και στις ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, και φυσικά να περιλαμβάνει τα διάφορα στοιχεία των ε, αντικειμένων του διαστήματος ώστε να αφυπνιστεί το κοινό και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάποιες εφαρμογές και για τις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιούμε τα... το two-line elements, το TLE των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι σημαντικό και χρήσιμο μοντέλο τις διπλές δηλαδή τροχιακές παραμέτρους των διαστημικών αντικειμένων. Η Αμέλεια προτείνει να συμπεριληφθεί και ο προπολογισμό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ε, κάτι που λέει στην τροπολογία 30 για το άρθρο 11. Δεν θα ήθελα να μείνει, δεν θα ήθελε η Αμέλεια να μείνει ο προπολογισμό μόνο στο παράρτημα και να προβλεφθεί η χρηματοδότηση από τις ε, πηγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ορίζον 2020, Γαλιλαίο, Κοπέρνικος, και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Βέβαια το θέμα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω με τους συναδέλφους και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ ότι πολύ σημαντικό σημείο για την εσωτερική ασφάλεια είναι να προστατευτούν οι ζωτική σημασία υποδομές. Οι υποδομές του διαστήματος και όλες οι σχετικές εφαρμογές που εξαρτώνται από αυτές τις υποδομές ε, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και ακόμη και αν δεν αναφέρεται επί χάρτου με σαφήνεια ε, το πόσο ζωτική σημασία είναι αυτές οι υποδομές του διαστήματος. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τον ε, προϋπολογισμό αυτό. Καταρχήν να το συμπεριλάβουμε στο νομοθετικό πλαίσιο και να δώσουμε ένα γενικό πεδίο εφαρμογή αλλά και ειδικού στόχους ήδη από το νομοθετικό κείμενο. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των διαστημικών μας υποδομών αυτό είναι ο απότερος στόχος του προγράμματος και θα πρέπει να το αναφέρουμε ήδη ε, στην πρόταση. Επίσης, θα πρέπει να προβλέψουμε μια δικτύωση των αισθητήρων για την επεξεργασία των δεδομένων και τις υπηρεσίε SST του άρθρου 3, επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, και να τις περιλάβουμε ως δράσεις και όχι ως στόχους ε, στο σημείο 19, που μιλά για τις ειδικέ δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πολιτές πρόγραμμα εργασίας. Ολοκληρώνει λοιπόν η Αμέλεια Αντερστότερ ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να εξετάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πριν τεθεί σε εφαρμογή με τη διαδικασία κατεξουσιοδότησης πράξεων του άρθρου 6. Αυτό αναφέρει ε, το σημείο 21 της έκθεσης. Και τέλος η Αμέλη σας ευχαριστεί για την προσοχή και συμφωνώ μαζί της. Σας ευχαριστώ και εγώ λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την συνάδελφο την κυρία Άντερς Στόντερ και τον εκπρόσωπό της. Η κυρία Κόβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ για το πρόγραμμα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος έχω να πω ότι όλοι μας εξαρτώμαστε από τις διαστημικές υποδομές. Διαφορετικά το κινητό τηλέφωνο δεν θα λειτουργούσε. Στο σχέδιο έκθεσης διευκρινίζονται από την εισηγήτρια κάποια πράγματα, κάτι που δεν συμβαίνει στο κείμενο της Επιτροπής. Ωστόσο πιστεύω ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη πρόοδο για το θέμα αυτό έτσι ώστε να έχουμε πραγματικές επιτυχίες. Για μένα προσωπικά τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα εξής. Καταρχάς η αβεβαιότητα του προϋπολογισμού. Η συγγήτρια προσέθεσε τα 70 εκατομμύρια στον ε, βασικό προϋπολογισμό. Εγώ όμως δεν είδα κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό αυτό. Υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα για το πρόγραμμα αυτό και αυτό με ανησυχεί. Ακόμα και αν ε, ορίσουμε ένα ακριβές ποσό στον προϋπολογισμό, ακόμα μου φαίνεται αβέβαιη η κατάσταση με το πρόγραμμα Κοπέρνικους και κινδυνεύουμε να μην ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Από την άλλη, πρέπει να δράσουμε ταχύτατα εντός αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ή δυνατόν πριν το τέλος της. Ακόμα και αν φανεί ότι βιαζόμαστε υπερβολικά. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Καλβάριο, είναι εισηγητής για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και πιστεύω πως πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την γνωμοδότηση αυτή πριν την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ε, το ζήτημα της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες έρευνας που συνδέονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτον, οι δράσεις του προγράμματος. Η συγκήτρια άλλαξε τη δομή δημιουργώντας ε, στόχους. Πιστεύω πως ε, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό που θα έχει το πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες δράσεις. Χρειάζεται βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής κάνοντας τη πιο συγκεκριμένη. Συνειδητοποιώ ότι θα είναι δύσκολο ειδικά θα είναι δύσκολο στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο προτιμά να παραμένει αόριστο. Χρειάζεται όμω να πιέσουμε από την αρχή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλο. Επίση, είναι θέμα του εάν τα κράτη-μέλη θα, είναι, θα συμμετέχουν σε, αυτό, σε αυτή τη σύμπραξη. Και πιστεύω πως δεν πρέπει να κλείσουμε πόρτες ε, στο θέμα αυτό. Αυτά πιστεύω ήταν τα κυριότερα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και πιστεύω επίσης ότι ο τρόπος ε, που ε, διαχειριζόμαστε την πρόταση, ο τρόπος που προτείνεται από την έκθεση είναι κάτι που χρήζει συζήτησης. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε δημιουργική συζήτηση στο μέλλον και σας καλώ να στηρίξετε τις τροπολογίες μου. Και πιστεύω και ελπίζω μάλλον η 7η Νοεμβρίου να εξακολουθεί να ισχύει ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ. Το, λόγο τον έχει ο συνάδελφος Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρα. Πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το πρόγραμμα της, ε, τοποθέτη, ε, του εντοπισμού των ε, αντικειμένων σε τροχιά είναι, πολύ, είναι ένα πρόγραμμα ε, κρίσιμο και πολύ σημαντικό για την διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στην ε, πολιτική του διαστήματος. Θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσει, να ανταγωνιστεί τις, ΗΠΑ τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τομέα ε, καινοτόμο της έρευνας και της ανάπτυξης με συνέπειες στην βιομηχανία μας και να μας επέτρεψε να μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις για τις διατλαντικές συμφωνίες με έναν μεγαλύτερο ρόλο και να υποστηρίξουμε την απασχόληση σε ένα τομέα ειδικής ή υψηλής εξειδίκευσης. συντήρηση και ο έλεγχος των όσων ε, συμβαίνουν στο διάστημα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ε, προσοχή που δείχνουμε σε όσα ε, ε, συμβαίνουν ε, στο έδαφος γιατί θα αποτελέσουν ουσιαστικά την σκηνή για, την, για μεγαλύτερη πολιτική σημασία στο μέλλον. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Στην αρχή είχαμε πει ότι η δημοσιονομική κάλυψη θα εξασφαλιστεί από τον, από τον, το, ορίζοντα, από το πρόγραμμα Horizon 2020 μετά από το Γαλιλαίο τώρα από το Κοπέρνικος, αλλά δεν είναι σαφές ε, ποια, ε, αν αυτή η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί και με ποιους πόρους. Γι' αυτό καλά έκανε και η συγγήτρια που ε, διευκρινίζει την, με οριστικό τρόπο ότι πρόκειται για 70 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο είναι αμεληταίο σε σχέση με τα τεράστια ποσά για τα οποία συζητάμε γενικότερα. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ε, υποβληθούν κάποιες τροπολογίες και θα υποβάλω τροπολογίες που θα καθορίσουν τον ρόλο ε, των ε, ασφαλιστικών εταιριών που συνήθως καλύπτουν τον κίνδυνο για τις πτήσεις στο διάστημα. Και θα μπορούσαμε να καλύψουμε επίσης και κινδύνους άλλου τύπου, παραδείγματος χάρη οι ηλιακές καταιγίδες. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω και τον, την δυνατότητα να υιοθετηθούν μέτρα για τον εντοπισμό με οπτικά μέσα και τηλεσκόπια, διότι θα επέτρεπαν να εντοπίσουμε και αντικείμενα ακόμα πιο μακρινά, διότι ο εντοπισμός με τα ραντάρ γίνεται πολύ πιο έντονος από την απόσταση. Επίσης δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να είναι το ο ρόλος που θα έπρεπε να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί μέσα στα πλαίσια όλου του διαστημικού, των άλλων, των άλλων διαστημικών προγραμμάτων, ίσως να δημιουργηθεί και κάποια ομάδα ad hoc υψηλού επίπεδου, που θα καθορίσει τις ε, περίπλοκες, αν θέλετε, σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για τα επόμενα 25 χρόνια. Επίσης και ένας ενεργός ρόλος της ΕΝΙΖΑ, που είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την προστασία των δικτύων και των πληροφοριών και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, διότι η πτυχή της ασφάλειας που δεν είναι και μόνο ε, θέμα ε, πληρότητας των δεδομένων ε, πρέπει να ε, υπογραμμιστεί με διαφορετικό τρόπο στο πρόγραμμα. Ευχαριστά, ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώχανσον θέλει να πάρει το λόγο. Γκλάντε. Κύριος Γκλάντε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, θα συμπληρώσω απλά αυτά που είπε ο συνάδελφο Πρόντι. Έχω και εγώ τι ίδιε αμφιβολίε σχετικά με τη χρηματοδότηση. Βρισκόμαστε εδώ ε, ε, σε μια περίπτωση που έχουμε μια υποδομή με το Γαλιλαίο, με το Κοπέρνικος, με το Έγνος και αυτή την υποδομή πρέπει να την προστατεύσουμε. Αν πάρουμε τώρα τα κονδύλια από αυτό το πρόγραμμα και τα διοχετεύσουμε αλλού, κινδυνεύουν τα εφιστάμενα προγράμματα. Ξέρω πως είναι λίγο περίεργο να δείχνει ένας ευρωβουλευτής ε, ε, πως συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πραγματικά εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά στοιχεία. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τον ε, προπολογισμό για τον ορίζοντα 2020, υπάρχουν πολλά ασαφή σημεία και πιστεύω πως πρέπει να δείξουμε ευελιξία. Έπειτα, με τις τεχνολογίες που διαθέτουμε και με τα μέσα που διαθέτουμε, πιστεύω πως ε, χρειαζόμαστε και περισσότερη έρευνα. Δεν αρκούν μόνο αυτά. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι δορυφόροι όσον αφορά τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκτόξευση πυράβλων, κατευθύνση πυράβλων κτλ. Όμως ε, υπάρχουν και κίνδυνοι όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία μετακινούνται αυτά τα αντικείμενα στο διάστημα. Και εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι η χρήση του προγράμματος ε, ορίζοντας 2020 είναι χρήσιμη. Ωστόσο, πρέπει να δείξουμε προσοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά το μέλλον, ε, διότι πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι το μέλλον των προγραμμάτων ε, που ε, τρέχουν και πιστεύω πως ε, πρέπει να ασχοληθούμε σε αυτή την νομοθετική περίοδο με διάφορα εκκρεμιστήματα, όπως για παράδειγμα την περίπτωση των ε, θραυσμάτων, των διαστημικών ε, σκουπιδιών, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν επιζήμια για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τις επικοινωνίες. Πάντως εντός της προθεσμίας θα υποβάλω και εγώ τις θετικές μου τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι συγγήτρια για τον προϋπολογισμό για το θέμα του συστήματος SST, επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος. Και γι' αυτό έχω καταθέσει και δύο τροπολογίες στην άλλη επιτροπή, στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα την καταθέσω και εδώ στην Ήτρε. Η μία τροπολογία εκφράζει τη λύπη της γιατί δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικό κείμενο προπολογισμό. Γι' αυτό θα ήθελα αυτά τα 70 εκατομμύρια να περιληφθούν και στο νομοθετικό κείμενο κατανεμημένα στην επταετία για το πρόγραμμα επιτήρησης και παρακολούθηση του διαστήματος. Επίση, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια από πού θα προέλθουν αυτά τα 70 εκατομμύρια, Ποιε θα είναι οι πηγέ χρηματοδότηση. Γι' αυτό και καταθέτω τροπολογία που λέει ότι και το Καλλιλέο και το Κοπέρνικους θα πρέπει να αποτελέσουν τι βασικέ πηγέ χρηματοδότηση για το πρόγραμμα SST. Ενώ ένα άλλο σύστημα, όπω και το Ταμείο εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να συμβάλλουν εφόσον καλύπτουμε και πτυχέ ασφάλεια. Και το πρόγραμμα Horizon 2020 θα πρέπει να συμβάλλει μόνο σε θέματα έρευνας. Ε, θέματα έρευνας του διαστήματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ορίζον 2020, αλλά μόνο και αυστηρά τα θεσιτήματα έρευνας. Αυτά ευχαριστώ. Bene. La Commission... Ωραία. Η Κομισιόν θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιό δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο στο στάδιο αυτό, όμως μία παρατήρηση θα θέλαμε να κάνουμε. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν αντικατοπτρίζουν την ανησυχία όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος. Η Κομισιόν διαρωτάται κατά πόσον η αναφορά σε ένα μέγιστο θα, μήπως θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση και με μια ελάχιστη συνεισφορά. Η μέγιστη συνεισφορά και η ελάχιστη συνεισφορά, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε την, το πρόγραμμα, τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Μία παρατήρηση μόνο, δηλαδή, αυτή την παρατήρηση θέλω να ε, κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Για τα συμπεράσματα, ο κύριος Γιώχανσον έχει το λόγο. Να πω εξ ονόματος της Αμέλεια, ε, ευχαριστώ για τα σχόλια και μια και δεν ήταν εδώ να τα ακούσει, θα τα πάρει γραπτά και θα τα σχολιάσει. Όμως σαν σκιώδης της Άλντε ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η συζήτηση για την ε, χρηματοδότηση. Και σαν αμέλεια να σας πω ότι θα είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στη συζήτηση με τους κοιόδης ε, και θα κάνει μια συζήτηση έτσι ώστε να βρεθεί ε, μια λύση. Λοιπόν, εκ μέρους της αμήλειας σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Γιώχανσον. Η προθεσμία την υποβολή των απολογιών είναι 13 Νοεμβρίου την ε, Τετάρτη. Μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. 7 Νοεμβρίου 2013 είναι η επόμενη συνεδρίασή μας από τις 9 στις 12.30. Είναι μια κοινή ε, ε, συνάντηση ένδυ και Ήτρε. Ενώ η επόμενη κανονική μας συνεδρίαση θα είναι 27 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Τελειώσαμε πιο γρήγορα. Έχετε κερδίσει και μία ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδήν.